Όποτε αποκατασταθούν οι προϋποθέσεις και οι όροι ασφάλειας, θα συνεχίσουμε τα σχέδια που έχουν διακόπτει προς το παρόν στο Βόρειο Μαλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Έχουμε 7 ψηφίσματα από την ECR, την EFD, τους πράσινους. Έκλεισε όμως η συζήτηση και στο τέλος θα γίνει η ψηφοφορία. Στη επόμενη περίπτωση αναφέρεται σε περιπτώσεις ατιμορρησίας στις Φιλιππίνες και καταρχήν θα μιλήσουν οι συντάκτες και ξεκινάει ο κύριος Δανέτσχη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι. Για μία ακόμη φορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναγκάζεται να υψώσει τη φωνή του ζητώντας σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην περιοχή αυτή της Ασίας και στη συγκεκριμένη χώρα τις Φιλιππίνες. Αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση επαναλαμβάνεται, δυστυχώς. Άρα μπορεί να μην είμαστε ανήμποροι, γιατί αν μη τι άλλο έχουμε το δικαίωμα να μιλήσουμε και να καταγγείλουμε τέτοιες καταστάσεις. Όπως είπε και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, χάρη στις προσπάθειές μας είχαμε κάποιες θετικές εξελίξεις στην Αίγυπτο. Θα πρέπει λοιπόν ε, να τελεσφορήσουν και οι προσπάθειές μας για τις Φιλιππίνες, γιατί η κατάσταση εκεί πραγματικά είναι απαράδεκτη. Έχουμε ε, καταστρατήγηση των ανθρωπιστικών ε, προδιαγραφών, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είναι αδύνατον να σιωπαίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ζανέτσκι. Για δύο λεπτά τώρα ο κύριος Ρωμέβα Ιρουέβα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός ότι οι εξοδικαστικές ε, ε εξοδικαστική έχουν σταματήσει εδώ και δύο χρόνια αλλά η δυνατότητα της κυβερνήσεως να πατάξει την ατιμορρησία δεν έχει προχωρήσει και αποδώσει και τελευταίως ε, είδαμε ότι ε, τα ε, ε, ε, οι μάρτυρες εις την δική και η πρόεδρος εκείνο εμπλέκονται και ε, δεν μπόρεσαν να μειωθούν οι δολοφονίες αλλά όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να μπορέσουμε όντως να προστατεύσουμε τον πληθυσμό διότι υπάρχουν πολλοί υποπτοί οι οποίοι είναι υπό αστυνομική παρακολούθηση χωρίς όμως να μπορεί να παταχθεί η βία ε, η οποία ε, απαιτεί την εφαρμογή της νομοθεσίας η οποία θεσπίστηκε το 2009. Θα πρέπει να υπάρχει μία αποζημίωση των θυμάτων και ζητούμε να υπάρχει ε, δράση της κυβέρνησης κατά τρόπον ώστε να διαλυθούν οι παραστρατιωτικές δυνάμεις και ζητούμε από την κυβέρνηση να ανακαλέσει ε, την απόφαση 546 ε, ε, ε, διότι απαιτούμε αυτά τα πράγματα εδώ και χρόνια και ακόμη δεν είναι δυνατόν να εισακουστούμε ίσως είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση και στα επόμενα έτη Ευχαριστώ κύριε Ρωμέβα Ρουέντα Κυρία Γιούλαντς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονό ότι τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί η ένταση της πολιτικής βία στην ε, ε, Φιλιππίνες. Αλλά παρόλα αυτά τα θύματα της σφαγής του Μαγκουιντανάου ε, δεν έχουν ακόμα δικαιωθεί. Ε, και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές περιπτώσεις βίων και ακούσεων εξαφανίσεων. Ε, η Πρόεδρος Ακίνο έχει δεσμευτεί για ε, καταπολέμηση της διαφθοράς και διάφορες άλλες βελτιώσεις οι οποίες προσπαθεί να εφαρμόσει. Ζητούμε από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να λάβει συγκεκριμένα μέτρα έτσι ώστε να προστατεύσει τους μάρτυρες σε δίκες, κυρίως δε όταν πρόκειται για δημοσιογράφους ε, και άλλα δημόσια ε, πρόσωπα. Ε, θα πρέπει οποιοδήποτε συλλαμβάνονται ως ύποπτοι για βίες ακούσεις εξαφανίσεις καθώς επίσης και για βασανιστήρια να συλλαμβάνονται άμεσα και να οδηγούνται ενώπιον των δικαστηρίων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό ο κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, έχουμε 72 ιδιωτικούς στρατούς και θεωρούμε ότι αυτή η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Ήδη όταν δημοκρατικά καράτη λειτουργούν με καταδίκες θάνατων θάνατον είναι απαράδεκτο αλλά οι ιδιωτικοί στρατοί πρέπει να καταπολεμηθούν. Αναγνωρίζουμε τις προσπάθειες της κυβερνήσεως Ακίνο οι οποίες είναι αξιέπαινες και προσπαθούν να προχωρήσουν αλλά πρέπει να εντείνουμε τα προγράμματα διότι ε, ε, στους ιδιωτικούς αυτούς στρατούς εμπλέκονται και οι μυστικές υπηρεσίες ε, και το παρακράτος και πρέπει η χώρα αυτή σιγά σιγά να μπορέσει να επανέλθει στην ένομο τάξη διότι είναι μια πλούσια και ωραία χώρα χώρα ένας βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρξει και να επικρατήσει κράτος δικαίου. Ευχαριστώ η κυρία Βερζιά για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στις Φιλιππίνες οι μη κυβερνητικές οργανώσεις εξακολουθούν να αναφέρουν ε, περιπτώσεις ε, βίων εξαφανίσεων, βασανισμών, ε, εξαφανίσεων ατόμων, κυρίως στρατευμένων της αριστεράς και δημοσιογράφων, καθώς επίσης και δολοφονίες. Βεβαίως ο αριθμός των δολοφονιών μειώνει, μειώνεται, αλλά παρόλα αυτά είναι η χώρα στην οποία από όλο τον κόσμο βλέπουμε τις περισσότερες περιπτώσεις εξαφάνισης και κακής μεταχείρισης των ανθρώπων του τύπου η ε, ε, ε, δίκη τη σφαγής του Μαγκουλιανάου όπου ε, σφαγιά περισσότεροι από 30 δημοσιογράφοι έχει ξεκινήσει αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Ε, πάντως ε, είναι κάτι θετικό αλλά βεβαίως δεν βλέπουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και η προστασία των, των μαρτύρων φαίνεται ότι είναι απλά λόγια όπως άλλωστε αποδεικνύει και ο φρικτός θάνατος του Ισμαήλ Αμίλ Ενόγκ τον οποίων ε, ε, σφαγίασαν ε, με πριόνι. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να ληφθούν νέα μέτρα. 4 με 10 εκατομμύρια ευρώ δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι ώστε να βελτιωθεί το δικαστικό σύστημα και η απόδοση της δικαιοσύνης έτσι ώστε να εξαφανιστούν οι εξωδικαϊκές διευθετήσεις και οι βίες εξαφανίσεις. Ελπίζω να εφαρμοστεί σωστά το πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τους συντάκτες ολοκληρώσαμε και ξεκινούν τώρα οι επόμενοι ομιλητές ξεκινώντας από τον κύριο Πρέντα. Ευχαριστώ. Λυπούμε για την δολοφονία των ε, ε, των ε, μαρτύρων στην περίπτωση του Μακιντανάου διότι είναι προφανές ότι η κυβέρνηση των Φιλιππινών πρέπει να συλλάβει τους υπευθύνου και αυτό το έγκλημα και να τους καταδικάσει. Θα πρέπει δε η δικαιοσύνη να μπορέσει να λειτουργήσει. Θέλω να σας υπενθυμίσω της όπως άλλωστε είπε και κάποιος συνάδελφος η δολοφονία τόσων ε, ε, δημοσιογράφων τα τελευταία χρόνια και ε, πέραν αυτών οι οποίοι τραυματίστηκαν ή διώχθηκαν διότι προσπάθησαν να κάνουν τη δουλειά τους και θα πρέπει να προσπαθήσουν με να προχωρήσουμε επιπλέον θα πρέπει να καταπολεμηθεί η διαφθορά η οποία επιτρέπει στην οικογένεια Μακτουά να λειτουργήσει με ατιμορρησία. Ευχαριστώ. Ε, η κυρία Κρετού για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η συζήτηση ε, έγινε ενώ ε, υπήρξε και άλλο ένα θύμα στην του μακελίου αυτού. 58 ε, άνθρωποι, μεταξύ άλλων γυναίκες και δημοσιογράφοι, έχασαν τη ζωή τους. Δεν μπορεί να συνεχιστεί ε, αυτή η ατιμορρησία στις Φιλιππίνες, γιατί απόρριά της είναι νέες δολοφονίες. Πολιτικές δολοφονίες και απαγωγές είναι πια καθημερινότητα στις ε, Φιλιππίνες και οι φυσικοί ευθουργοί ενθαρρύνονται από την προστασία που τους παρέχει η η μη ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Επίσης, δημοσιογράφοι δέχονται απειλέ κατά τη ζωή τους, υφίστανται παρενόχληση και μερικές φορές χάνουν και την ίδια τους τη ζωή. Γίνονται διάφορες συγκρούσεις μεταξύ των τοπικών φατριών και δυστυχώς επιτείνεται η αρνητική πολιτική κατάσταση, η έλλειψη δημοκρατίας και οι φτώχεια Φιλιππίνες. Θα πρέπει η κυβέρνηση να αντιδράσει στα μέτρα, στην κατάσταση αυτή και να λάβει κάποια μέτρα για να αποκαταστήσει, να αποκαταστήσει το κράτος δικαίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κρέτσου. Η κυρία Σάκη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Ο πρόεδρο εκείνη είπε ότι ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η χρηστή διακυβέρνηση και η καταπολέμηση τη διαφθορά ήταν ε, προτεραιότητα. Θέλει να περιοριστούν οι εξοδικαστικέ εκτελέσει και άλλε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η δήλωση ήταν πολύ θετική και χαίρομαι για την έγκριση του καταστατικού, για το, του καταστατικού της Ρώμης από τις Φιλιππίνες. Αλλά τώρα πρέπει από τα λόγια να περάσουμε στα έργα. Πολλοί είναι οι λόγοι ανησυχίας για την ατιμορρησία στις Φιλιππίνες. Ε, δολοφονούνται μάρτυρες, ε, δημοσιογράφοι είναι από τις πιο επικίνδυνες χώρες ε, για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρειάζονται κατεπηγόντως μέτρα για να προστατευτούν μάρτυρες, εισαγγελείς, ανακριτές, δημοσιογράφοι που εμπλέκονται σε ευαίσθητες δίκες. Θα πρέπει να σταλεί μήνυμα ότι θα σταματήσει η τιμωρησία για τις εξοδικαστικέ δολοφονίες, αναγκαστικές εξαφανίσεις και τα βασανιστήρια και θα προσάγονται στην δικαιοσύνη οι υπέτειοι, ακόμη και αν είναι υψηλά ιστάμενοι ή έχουν υψηλές θέσεις σε στρατιωτικές ή παραστρατητικέ δομές. Ε, καλό θα ήταν να επισκεφθεί και ο ειδικό απεσταλμένο στο ΙΕ τη χώρα αυτή για να ελέγξει την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και φυσικά θα πρέπει να βοηθήσουμε το πρόγραμμα Δικαιοσύνη για Όλου, που είναι πρικοδοτημένο με 10 εκατομμύρια ευρώ ε, μέχρι το 2015, 2012 με 2015. Ο κύριος Πάσκα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, υπάρχει μια τραγική κατάσταση η οποία συνεχίζεται στις ε, Φιλιππίνες με εμπλοκή ιδιωτικών στρατών, του κρατικού στρατού και της κυβερνήσεως. Αλλά θα χρειαστεί να συνεργαστούμε με, τα, με τους κρατικούς οργανισμούς για να βρεθεί μία διέξοδο από την κατάσταση αυτή. Δεν είναι δυνατόν σε έναν πολιτισμένο κόσμο το κράτος να επιτρέπει ε, να ε, καλύπτουν το έργο της ασφαλείας ιδιωτική στρατή ε, για τους οποίους δεν ευθύνεται το κράτος αλλά το, η κυβέρνηση είναι η υπόλογη και δεν μπορούμε να δεχθούμε πλέον αυτή τη συμπεριφορά της κυρίας Ακίνο. Θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της η κυβέρνηση της, των Φιλιππινών και να μην επιτρέψει να συνεχίζεται αυτές οι εξοδικαστικές δράσεις. Ευχαριστώ. Ολοκληρώθηκαν οι ομιλίες των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων και τώρα πρώτος ο κύριος Κέλλη. Όπως υπόθηκε ήδη, η κατάσταση στις φιλεπίδες δεν είναι καθόλου ευχάριστη και ούτε είναι άλλωστε η πρώτη φορά που τη συζητάμε εδώ στο Κοινοβούλιο. Οπωσδήποτε αυτές οι σφαγές ε, ε, ειδικά μεταξύ του 9 και του 11 ε, όπου δολοφονήθηκαν πάνω από 57 δημοσιογράφοι είναι απαράδεκτες και η έλλειψη καταδικών όσον αφορά τους υπευθύνους μας απασχολεί ιδιαίτερος. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο μετά την, από τη στιγμή που η πρόεδρος Ακίνο ανέλευε την εξουσία βλέπουμε ότι υπάρχει σαφής μείωση της βία. Ε, βίας. Όμως θα πρέπει και η πρόεδρος Ακίνο να πάρει ε, συγκεκριμένα μέτρα. Βλέπουμε κάποια βελτίωση αλλά δεν αρκεί. Θα πρέπει να ε, ασκηθούν πιέσεις έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον ατιμορρησία για όσους έχουν ασκήσει βία είτε είναι της αστυνομίας είτε είναι του στρατού κλπ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Τώρα ακολουθεί η κυρία Κέντιγκεν Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι διοκτικέ αρχέ και η δικαιοσύνη στι Φιλιππίνες δεν λειτουργούν σωστά, κάτι που επιβεβαιώνει και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στα συμπεράσματα του Μαΐου. Επιπλέον, το επίπεδο βία κατά των δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων έχει ε, ε, αυξηθεί αισθητά από την προηγούμενη έκθεση του 2008. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη, τα γεγονότα του 2009 όταν ένοπλοι άνδρες από τη φατρία Πατουάν με τη βοήθεια της τοπικής αστυνομίας έστησαν ενέδρα ε, σε πολίτες που υποστήριζαν τον ε, υποψήφιο της αντιπολίτευσης για τις, εκλογές, ε, για τις τοπικές εκλογές. Και μάλιστα, ω συνέπεια αυτή τη βάναυση επίθεση, 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή του, μεταξύ των οποίων και ξένοι δημοσιογράφοι. Η δικαιοσύνη σκεμμένα κολλησιέργησε και τα αποτελέσματά τη ούτω ή άλλω ήταν αποτελεσματικά. Η έλλειψη αποτελεσματικότητα και ε, διαφάνεια των διοκτικών αρχών δημιουργεί σοβαρέ ανησυχίε για την ανεξαρτησία του. Δεν θα πρέπει να παραμείνουν τιμώρητε αυτές οι παράνομε εκτελέσεις και οι απαγωγέ. Θα πρέπει επιτέλους να εξασφαλίσει ε, επαναφορά του κράτου δικαίου στην χώρα η κυβέρνηση των Φιλιππινών. Ευχαριστώ για ένα λεπτό ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. από την ε, βία, τις βίες ε, δολοφονίες 8 ατόμων στην επαρχία Βογγεντενάου βλέπουμε ότι οι υπεύθυνοι ακόμη έχουν εξέχουσες θέσεις εις ε, την περιοχή και διατηρούν ε, ε, ιδιωτικούς στρατούς. Η τραγωδία του Μαγκιντανάου και ε, οι επιπτώσεις της αποδεικνύουν ότι η χώρα αυτή έχει εγκαταλείψει οποιοδήποτε ίχνος δημοκρατίας και μπαίνει προς το χάος. Γι' αυτό και πρέπει να απαγορευτούν αμέσως όλη η στρατή αυτή και να τιμωρηθούν οι πέτειες ε, μέσω δικαστικών διαδικασιών. Ευχαριστώ κύριε Παλέτσκης. Έτσι έληξε ο κατάλογος των ομιλητών. Ερχόμαστε τώρα στη διαδικασία Catch the και δίνω πρώτα τον λόγο στον κύριο Σιλβέστρης. Η σφαγή του που έλαβε χρόνο το 2009 ε, ε, και είχε είχε σαν θύματα 58 ε, ανθρώπους ενώ οι δημοσιογράφοι οι δικηγόροι, οι οδηγοί πήγαιναν σε αυτήν την πόλη έτσι ώστε να υποβάλουν την υποψηφιότητα του δημάρχου του οποίου η γυναίκα επίσης έχασε τη ζωή του εκεί. Ε, έχουμε 25 ε, θανατικές ε, πίνες για τον Αντάλ Αμπατουάν ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε δίκη για σφαγή και τα λοιπά αλλά πρόκειται για μια οικογένεια πάρα πολύ δυνατή οπότε είναι λίγη λίγοι οι μάρτυρες οι οποίοι φτάνουν στο δικαστήριο για να γίνουν μάρτυρες κατηγορίες. Ε, θα πρέπει οπωσδήποτε οι Φιλιππίνες, η κυβέρνηση των Φιλιππίνων να κυρώσουν τις διεθνείς συμβάσεις για την προστασία των ατόμων, από οποίες εξαφανίσεις κλπ. Ε, και να πάρουν συγκεκριμένα μέτρα. Ευχαριστώ κύριο Στρέπο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η ατιμορρησία και η διαφθορά είναι όλο και γίνονται όλο και μεγαλύτερη μάστιγα στις Φιλιππίνες. Τα προβλήματα της θεωροδοκίας και της διαφθοράς ε, απομάκρυναν τους ε, επίδοξους επενδυτές από τις Φιλιππίνες. Είχαμε και τη σφαγή του Μακινταναό το 2009. Οι μάρτυρες του μακελιού αυτού δολοφονήθηκαν. Αυτό είναι επέσχυντο για την ε, φιλιππινέζικη δικαιοσύνη. έχουμε και υποχρεωτικές αναγκαστικές εξαφανίσεις ε, με πολιτικά κίνητρα. Οι Φιλιππίνες θα πρέπει να, να, να τηρήσουν τις διεθνείς τους δεσμεύσεις και να προστατεύουν τους μάρτυρες και τις οικογένειές τους. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυ εξελίξεις της πολιτικής κατάστασης της Φιλιππίνες και κυρίως ε, τη διεξαγωγή της δίκης για το μακελιό του Μακίντα Ναό. Ευχαριστώ κύριο Σταβάδε. Ευχαριστώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητούμε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την περίπτωση του μακελιού του Μακιντανάου. στι αρχέ του 2010 είχαμε συντάξει σχετικό ψήφισμα για τη σφαγή εκείνη, που, ε, όπου έχασαν τη ζωή τους περίπου 100 άτομα σε ένα νησί των Φιλιππίνων, ε, Φιλιππίνων και μάλιστα 30 από αυτού ήταν και δημοσιογράφοι. Αυτό έγινε το 2010. Το 2011 ε, παρόλο που συγκεντρώθηκαν ε, πάρα πολλές ε, μαρτυρίες και καταθέσεις, από ό,τι φαίνεται από τους δικηγόρους των θυμάτων, η, η, η δικαιοσύνη κολυσιεργεί. Βέβαια, ελπίζουμε να τηρήσει τις διακηρύξεις του πρόεδρος της της χώρας αυτής και να τηρηθούν οι διεθνείς δεσμεύσεις, να γίνει δίκαιη δίκη και μάλιστα να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για μια τέτοια δίκαιη δίκη. Αλλιώς να ζητήσουν οι Φιλιππίνες διεθνή, ε, διεθνή βοήθεια. Θα, πάνω από 70 είναι οι ένοπλες παραστρατιωτικές δυνάμεις στις Φιλιππίνες. Αν είναι ανίκανη να τις εξαρθρώσει η κυβέρνηση θα πρέπει να ζητήσει τη διεθνή βοήθεια για να το κάνει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ταβάρες, ο κύριος Τάνοκ τώρα. Mm. Χωρίς μικρόφωνο. και εγώ θέλω να εκφράσω την ανησυχία μας για ε, το κράτος ατιμορρησίας που εξελίχθηκε τα τελευταία χρόνια στις Φιλιππίνες μετά την δολοφονία 57 ατόμων συμπεριλαμβανομένων και δημοσιογράφων που συμμετείχαν σε μια ειρηνική πορεία στο Μιντανάο. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ε, ευρεία διαφθορά ε, και τρομοκρατία και μοιάζει με την κατάσταση της Σομαλίας που καταπιέζει την ελευθερία. Γι' αυτό και παρακαλώ την πρόεδρο Ακίνο να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα του λαού της και να θεσπίσει ένα πρόγραμμα προστασίας των μαρτύρων και ε, ε, να ε, μην επιτρέψει στην αντιπολίτευση να λιμένεται τη χώρα που είναι τόσο ωραία. Ευχαριστώ. Και ολοκληρώνοντας τη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙ, η κυρία Κόρολα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτή η έλλειψη αποδόσης δικαιοσύνη και η ατιμορρησία ε, είναι ιδιαίτερα έντονη στις ε, Φιλιππίνες. Ε, έχουμε, έχουν βρεθεί ας πούμε σώματα ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί μετά από πάρα πολύ καιρό μετά την εξαφάνισή τους. Επίσης εξαφανίζονται μάρτυρες κυρίως της σφαγής του Μαγκεντανάου, έχουν ήδη θανατωθεί τρει. Πρόκειται επομένω για πραγματικές πολιτικές δολοφονίες. Έχουμε επίσης τουλάχιστον 7 περιπτώσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά σημαντικές και βεβαίως και μετά την εγκατάσταση της νέας κυβέρνησης εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα. Έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση στις Φιλιππίνες, αλλά παρόλα αυτά ε, το ε, ποινικό δικαστήριο των ε, Φιλιππίνων αποδεικνύει ότι δεν εφαρμόζει τελικά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Βλέπουμε ας πούμε τι έγινε και στα Ηνωμένα Έθνη για την Συρία, ενώ δεν έγινε για τις Φιλιππίνες Φιλιππίνες. Οπωσδήποτε θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να συνεχίσει ε, ε, ε, να δρά και όχι να περιμένει με σταυρωμένα τα χέρια. Ευχαριστώ πολύ. Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνω τον λόγο στον Επίτροπο κύριο Ντάλη. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου το ζήτημα της ε, ατιμορρησίας των εξοδικαστικών ε, ε, θανατώσεων και παραβιάσεων των δικαιωμάτων είναι δυστυχώς στοιχεία τα οποία γνωρίζουμε εδώ και καιρό και παληθεύονται στις Φιλιππίνες. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση βοηθάει την χώρα έτσι ώστε να εφαρμόσει πρόγραμμα στήριξης της δικαιοσύνης. Δύο εβδομάδες μόλις πριν η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μέσω των μελών ε, που, έχουν, που εδρεύουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας συζήτησαν το θέμα των ε, Φιλιππινών όσον αφορά και, και συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν την απόδοση δικαιοσύνης, την ατιμορρησία κλπ. Καλωσορίζω το γεγονός ότι με αυτή την ευκαιρία η κυβέρνηση των Φιλιππίνων ε, παρουσίασε ε, ε, πρόγραμμα για την εφαρμογή ε, της ε, προστασίας ε, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχει επίσης ξεκινήσει η Πρόεδρος Ακίνο από τη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία διεργασίες έτσι ώστε να απονεμηθεί γρηγορότερα η δικαιοσύνη όσον αφορά την, τους υπεύθυνους για τη σφαγή του Μουγκουιντανάου. έγιναν και άλλες προσπάθειες αντιμετώπισης ε, του προβλήματος ε, αλλά αυτή τη φορά πιστεύουμε ότι μέσω των δράσεων του Προέδρου Ακίνο πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση θα ε, οδηγούμεθα σε, σε καλό δρόμο όσον αφορά το τέλος ε, της, ε, της ατιμορρησίας. Επίσης ζητούμε από την κυβέρνηση των Φιλιππίνων να κυρώσει τη Διεθνή Σύμβαση για, την, για το κατά των βασανισμών και η αποδοχή από πλευράς κυβερνήσεως είναι κάτι θετικό εμείς ζητούμε και ενθαρρύνουμε την Πρόεδρο Ακίνο ε, όχι μονάχα να οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης όλους όσους παραβίασαν τα ανθρώπινα δικαιώματα ή ε, ε, τους νόμους σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα τα τελευταία χρόνια αλλά να σταματήσει γενικότερα η ατιμορρυσία στη χώρα. Είναι γεγονός ότι το πρόγραμμα EP-JUST έχει ήδη δώσει κάποια πρώτα καλά αποτελέσματα Είχαμε το 2006 ε, ε, ας πούμε 300 ε, περιπτώσεις εξοδικαστικών εκτελέσεων και ο αριθμός τους έχει πέσει πάρα πολύ τον τελευταίο χρόνο. Πρέπει να σας πω και να σας διασφαλίσω ότι εξακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεργάζεται στενά ε, με τις Φιλιππίνες όσον αφορά τον τομέα της ε, ε, δικαιοσύνης. Πρόσφατα έχουμε εγκρίνει ένα πρόγραμμα 10 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο εφαρμόζεται στα πλαίσια του EP Justa έτσι ώστε να βελτιωθεί η απόδοση, η απόδοση ποινικής δικαιοσύνης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Νταλή. Ε, έχουμε ε, επτά ψηφίσματα στο τέλος της συζητήσεως τα οποία θα ψηφιστούν στο τέλος. Μετά την επόμενη συζήτηση ακολουθεί